Ξέχασα την, ε, να ευχαριστήσω την κυρία Μπάσο και την κυρία Σαρτόρη όταν ανέφερα τη συνεργασία μου με του κοιόδη Μία από τι αδυναμίε που <laughs> υπήρχαν στην έκθεση και αυτή που ξέχασα να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι. Επόμενο θέμα, σύμφωνα με τη Μέση Διάταξη, είναι η ώρα των ερωτήσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρώτη ερώτηση είναι του κυρίου Παρνιό προς τον Επίτροπο κύριο Ντάλη και αφορά την απαγόρευση κυκλοφορίας του φαρμάκου Mediator. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε, όποτε θέλετε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ και ε, σε κάθε μία από τις τέσσερις ερωτήσεις ξεχωριστά. Η πρώτη ερώτηση ήταν, μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξηγήσει για ποιο λόγο δεν ελήφθη η απόφαση το 1998 να απαγορευτεί η κυκλοφορία ε, φαρμακευτικών προϊόντων που ε, περιέχουν την ουσία Benfluorex. Το 1998 συζητήθηκε αυτό στην αντίστοιχη επιτροπή, η οποία ονομάζεται τώρα Επιτροπή για Φάρμακα για ε, Ανθρώπινη Χρήση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και στη συνέχεια στην Ομάδα Εργασίας για τη Φαρμακοεπαγρύπνηση. Θεώρησε τότε η Επιτροπή ότι η ουσία Ben Fluorex δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο πεδίο ε, εφαρμογής και διαδικασίας μόνιμης αξιολόγησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως, ε, ε, κάποιους παράγοντες που ε, κόβουν την όρεξη ε, ωστόσο, συμφωνήθηκε η αντίστοιχη ομάδα εργασίας να διερευνήσει το θέμα αν υπήρχε ζήτημα ασφαλείας δηλαδή με την ουσία αυτή. Το Μάρτιο του 1999 η ομάδα εργασίας για τη φαρμακοεπαχρύπνηση κατέληξε ότι δεν υπήρχε ε, βασικός λόγος ανησυχίας ε, για ε, φάρμακα που περιλαμβάνουν την ουσία Benfluorex. Ε, στη συνέχεια η συζήτηση στην ομάδα εργασία δεν οδήγησε σε αλλαγέ στην απόφαση αυτή. Ερώτηση δεύτερη. Δεν θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είχε ειδοποιηθεί για πρώτη φορά από τις απαγορεύσεις που είχαν επιβληθεί στην Ισπανία και στη ε, Ιταλία. Απάντηση. Η Ιταλία και η Ισπανία δεν ανακάλεσαν την άδεια κυκλοφορίας ε, της ουσίας Ben Fluorex. Για πρώτη φορά ε, έλαβε πραγματικά μέτρα ένα κράτος για απόσυρση του Mediator το, ήταν το 2009 όταν η Γαλλία σταμάτησε, ε, απέσυρε την έγκριση και ε, κυκλο, άδεια κυκλοφορίας. Στην Ισπανία η Σερβιέ η ίδια η εταιρεία ε, η παρασκευάστρια το 2003 απέσυρε το φάρμακο χωρίς απαγόρευση. Η ίδια η Σερβιέ λοιπόν αντίστοιχα δεν ζήτησε ανανέωση της άδεια κυκλοφορίας το 2003 ε, στην Ιταλία. Παρέμεινε λοιπόν η κυκλοφορία το προϊόν στη ε, Γαλλία, Πορτογαλία, Λουξεμβούργο και στην Ελλάδα. Το Benfluorex συζητήθηκε στην ομάδα φάρμακο επαγρύπνησης που είναι και το φόρουμ για τα κράτη-μέλη για να ανταλλάσσουν στοιχεία φάρμακο επαγρύπνησης μεταξύ τους. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η παρακολούθηση των στοιχείων φάρμακο επαγρύπνησης και η επόμενη λήψη αποφάσεων για τις εθνικές άδειε κυκλοφορίας ιατρικών προϊόντων και φαρμάκων ε, παραμένει στα χέρια των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτάκτως επεμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις και ε, αυτό βλέπετε πολύ συγκεκριμένα από την νομοθεσία. Είναι πολύ περιορισμένες. Μπορεί να ζητήσει αξιολόγηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δύο περιπτώσεις. Πρώτον, όταν τα κράτη-μέλη έχουν ε, αποκλίνουσες αποφάσει ω προ την άδεια κυκλοφορία ενό φαρμάκου και δεύτερον, όταν ε, πρόκειται για αλλαγή, ανάκληση, διαφοροποίηση της άδειας κυκλοφορίας και ε, όταν μας ε, χρειάζεται φαρμακοεπραγρύπνηση και όταν θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι διακυβεύονται τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αποφάσισε η αντίστοιχη ομάδα εργασία. Δεν είχαμε αποκλίνουσε αποφάσει από τα κράτη-μέλη τα ίδια και ε, ούτε διαφορετική απάντηση στη συζήτηση της Φάρμακοεπαγρύπνησης. Η τρίτη ερώτηση, γιατί δεν έδρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2010 όταν λήφθη σαφή ε, απόφαση για την κυκλοφορία στην αγορά αυτή τη ουσία. Απάντηση. Το 2009 μόνο ένα κράτος μέλος η Γαλλία διέκοψε την κυκλοφορία ε, ε, της ε, ουσίας αυτής και του Μεντιατόρ από το 2004 και μετά ισχύει μια νομοθεσία που σημαίνει ότι αυτόματα δρομολογείται μια διαδικασία η οποία οδήγησε στη λήψη απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που καλεί όλα τα κράτη-μέλη ε, να αποσύρουν οποιασδήποτε άδειες κυκλοφορίας προϊόντων που περιέχουν τη δραστική ουσία Benfluorex. Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι η νέα νομοθεσία για τη φαρμακοεπαγρύπνηση που εγκρίθηκε στις 15 Δεκεμβρίου του 2010 εισαγάγει επιπλέον διατάξει ε, για να ε, υπάρχει ε, μια έγκαιρη προειδοποίηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ε, ως προς τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δημιουργούνται και νέες διαδικασίες εκτίμησης ε, της ασφάλειας τέτοιων προϊόντων ε, και αυτό οδηγεί σε εναρμονισμένη δράση των κρατών μελών. Τέταρτη και τελευταία ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απευθυνθεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και να ζητήσει μια πλήρη έρευνα αναδρομικά ε, για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε αυτό το φάρμακο επί μια εικοσαετία και πλέον. Απάντηση. Μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ζητήσει από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων να κάνει μια τέτοια πλήρη αναδρομική διερεύνηση της υπόθεσης και του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε πάνω από μία εικοσαετία το φάρμακο αυτό. Τα στοιχεία και η τεκμηρίωση που αναφέρονται στην γαλλική έκθεση δείχνουν σαφώς ότι ε, στη Γαλλία ήταν η μεγαλύτερη χρήση με μεγάλη διαφορά του φαρμάκου αυτού. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Να σας πω πώς θα χειριστώ απόψε τις συμπροματικές ερωτήσεις. Θα τις ομαδοποιώ θυμάστε ότι έχετε 30 δεύτερα ο καθένας για τη συμπληρωματική σας ερώτηση και μετά θα ζητήσω από τους επιτρόπους να απαντούν σε όλες τις συμπληρωματικές ε, ερωτήσεις μαζί. Παρακαλώ. Ο κύριος Παρνιό. Σύντομη συμπληρωματική ερώτηση μετά τις απαντήσεις που μας έδωσε ο Επίτροπος Δάλη. Καταρχήν ευχαριστώ θερμά τον Επίτροπο για την ε, ακρίβεια των απαντήσεών του και τη σχολαστικότητα. Διαπιστώνουμε, όπως είπατε και εσείς, ότι 2003 και 2005 το εργαστήριο Σερβιέ ζήτησε να μην ε, ανανεωθεί η άδεια και να μην κυκλοφορεί στις δύο χώρες αυτό το φάρμακο. Μεταξύ 98 ε, και 99 δεν είχε ζητηθεί καν η απαγόρευση κυκλοφορία του εγγράφου, ενώ γνωρίζουμε ότι το Mediator ήδη από το 1997 είχε απαγορευτεί στι Ηνωμένε Πολιτείε. Και μάλιστα σε μια τόσο σημαντική αγορά όπω είναι η ευρωπαϊκή αγορά, με 500 εκατομμύρια καταναλωτέ, διαπιστώνουμε και αυτή είναι η συμπληρωματική, του, η συμπληρωματική μου ερώτηση, είναι ότι απαιτείται μια ε, περαιτέρω επαγρύπνηση και κάποια προειδοποιητικά μηνύματα ώστε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε μια ισχυρή αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και να αποφεύγουμε αυτό που συνέβη σε πολλές χώρες μέλη με... και να μην επαναληφθεί αυτό που συνέβη στη Γαλλία. Επαναλαμβάνω ότι οι συμπληρωματικές ερωτήσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν το μισό λεπτό. Αυτό προβλέπουν οι κανόνες και έχουμε πολλές συμπληρωματικές ερωτήσεις και θέλω να ολοκληρώσουμε το απόγευμα της ερωτής προς την Επιτροπή. Η επόμενη ερώτηση είναι του κυρίου Ταραμπέλα. Κύριε Επίτροπε, ας διευρύνουμε τη συζήτηση γιατί το θέμα του Μεδιάτορ είναι η ορατή κορυφή μόνο του παγόβουνου. Γιατί ένα φάρμακο που μπορεί να θεωρείται επικίνδυνο ή και μοιραίο, ενώ αποσύρεται από την αγορά σε ορισμένε χώρε, μπορεί ελεύθερα να κυκλοφορεί στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να σκεφτούμε το ρόλο και την αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, γιατί τα συμπεράσματα του δεν είναι αποτελεσ... δεσμευτικά, υποχρεωτικά για τα κράτη-μέλη. Ο επίτροπο. οι διαδικασίες που ίσχυαν κατά τη διάρκεια των ετών αυτών που έλαβαν χώρα τα πραγματικά περιστατικά που σας εξιστόρισα προέβλεπαν ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής ε, Αρχής. Και μάλιστα αυτή, αυτός ο διαχωρισμός εξακολουθεί να ισχύει τα κράτη-μέλη επιμένουν σε αυτό. Γι' αυτό και σκεφτήκαμε ότι μου ήταν να ενισχύσουμε τις διαδικασίες μας για την φαρμακο Και μάλιστα το 2004 είχαμε μια σημαντική πρόοδο με την αναθεώρηση των διαδικασιών φάρμακοεπαγρύπνησης. Και μάλιστα στην τελευταία συμφωνία φάρμακοεπαγρύπνησης, αυτή που ισχύει τώρα, έχουμε πολλές δράσεις ε, που μπορούν να αναλυφθούν, να αναλυφθούν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε οποιαδήποτε ουσία ή φάρμακο που αποσύρεται από μία αγορά να κυκλοφορεί αυτός πληροφορία και να λαμβάνεται μία απόφαση, κάτι που δεν γινόταν προηγουμένως. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. και έχω δώσει εντολές και στις υπηρεσίες μου να δοκιμάσουν τις νέες διαδικασίες φαρμακοεπαγρύπνησης, αυτές που θεσπίστηκαν μετά την τελευταία συμφωνία περί φαρμακοεπαγρύπνησης. Και μάλιστα το φάρμακο Mediator θα είναι μια περίπτωση αναφοράς, μια υπόθεση αναφοράς για να δούμε αν ίσχυαν οι τελευταίες, ε, τελευταίες διαδικασίες φαρμακοεπαγρύπνησης. Θα είχαμε αντίστοιχη περίπτωση με αυτή του Μεντιάτορ. Θέλουμε να αποφύγουμε στενοπούς, να αποφύγουμε προσκόμματα και να μην εμποδιστούμε στην ε, λήψη απόφαση. Αν διαπιστώσουμε τέτοια προβλήματα στη διαδικασία, θα προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε και θα σας ενημερώσουμε. Προχωράμε λοιπόν τώρα στην επόμενη ερώτηση από τον κύριο Μπέλετ ε, που απευθύνεται ε, στον Επίτροπο Πίτμπαξ ε, σας καλωσορίζουμε και αφορά στις συνδρομές iPad από την Apple. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, η ε, Apple, ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει ψηφιακές ε, συνδρομές ε, για τα περιοδικά μόνο μέσα από τις εφαρμογές που πολλούνται στα καταστήματά της online. Βεβαίως ε, αυτό ε, θα γίνεται μέσα από website ε, ή και με άλλες δυνατότητες, όμως δεν θα μπορούν να έχουν συνδρομές μέσω του iTunes. Τώρα, κατά πόσον η συμπεριφορά της Apple αποτελεί παραβίαση του κανονισμού ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό εξαρτάται βέβαια από οικονομικά και νομικά και άλλα στοιχεία. Η Apple έχει ίσως πράγματι δεσπόζουσα θέση στην ε, αγορά και τα όρια όμως της αγοράς αυτής ε, δεν είναι σαφή. Ε, ως τομέας είναι νέος και εξελίσσεται περαιτέρω. Επίσης ε, υπάρχουν και πολλές άλλες ε, συγκρίσιμες ε, πλατφόρμες και συσκευές που προσφέρουν παρεμφερείς λειτουργίες. Ορισμένες εξ αυτών στηρίζονται μόνο από καταστήματα online. Η ζήτηση των καταναλωτών για ηλεκτρονικές εφημερίδες δεν είναι σαφής, εξελίσσεται περαιτέρω. Από τη στιγμή λοιπόν που η αγορά θα είναι σαφώς εντοπιζόμενη, τότε θα πρέπει να εξολογηθεί το θέμα της δεσπόζουσας θέσης. Η δεσπόζουσα θέση ορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ως μια θέση οικονομικής ισχύω, την οποία απολαμβάνει μια επιχείρηση και αυτό της δίνει τη δυνατότητα να παρεμποδίζει τον ανταγωνισμό στη συγκεκριμένη αγορά η εταιρεία δηλαδή μπορεί σε μεγάλο βαθμό ε, να συμπεριφέρεται ανεξάρτητα από τους ε, πελάτες ε, και τους ανταγωνιστές και σε τελική ανάλυση από τους καταναλωτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει ότι υπάρχουν εναλλακτικέ πλατφόρμες και αρκετές εταιρείες πρόσφατα εισήγαγαν ή προβλέπεται στο εγγύς μέλλον να εισάγουν παρεμφερείς συσκευές από πλευράς λειτουργικότητας. Θα μοιάζουν από με το iPad. Έτσι λοιπόν η Επιτροπή ε, παρακολουθεί τις εξελίξεις όσον αφορά την εμπορική πολιτική της Apple, παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Πρόεδρος. Ε, και πάλι, όπως σας είπα, ε, θα εξτάσω από κοινού όλες τις συμπληρωματικές ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα δίνω το λόγο στον κύριο Μπέλετ. Ευχαριστώ. Γεια σας, εδώ είμαι. Η Apple είπε ότι θα δώσει ένα νέο μοντέλο ε, στους συνδρομητές, αλλά το θέμα είναι η δεσπόζουσα θέση. Κύριε Επίτροπε, ε, θέλει να ε, ελέγχει πληροφορίες και στοιχεία για τους πελάτες η Apple και αυτό είναι βλαβερό για το μέλλον της πληροφορικής στην Ευρώπη και για τον ανταγωνισμό. Αυτό είναι το θέμα, η δεσπόζουσα θέση και τι θα κάνετε ε, και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Είναι υπόθεση εβδομάδων, υπόθεση μηνών. Πότε προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Ζέμκα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την απάντησή του. Αλλά κατά τη γνώμη μου δημιούργησε κάποιο προβληματισμό και έγινε και πολύ θεμελιώδη ζητήματα. Έχουμε, μπορούμε να φανταστούμε τι μερίδιο της αγοράς μπορεί να κατακτήσει το νέο προϊόν της ε, Apple. Γιατί δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία ακόμη. Αλλά είναι μια πληροφορία που ε, χρειαζόμαστε γιατί υπάρχει σημαντική απειλή να δημιουργηθεί ε, δεσπόζουσα θέση της Apple ε, στην ευρωπαϊκή αγορά και κατάχρηση αυτής. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος. Θα το δούμε. Θα το δούμε αν ε, αποκτήσει δεσπόζουσα θέση Apple στην αγορά, γιατί είναι μια αγορά εν εξελίξη. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις ε, μελέτες, την αξιολόγηση, ποια είναι αυτή η αγορά, τι διαστάσεις έχει και τι τη δεσπόζουσα θέση σε μια τέτοια αγορά. Αλλά η αγορά αυτή βρίσκεται στα σπάργανα, είναι ακόμη μικρή, δεν ε, έχει νόημα. Είναι πολύ πρόημο να μιλήσουμε για οποιαδήποτε δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν υπάρχουν ε, ανταγωνιστικές προτάσεις ε, και η απάντηση της Apple δεν ε, στοιχειοθετεί πόσο θέση, δεν, υπάρχει, δεν έχει νόημα να αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακολουθούμε την κατάσταση ε, και την τήρηση των ευρωπαϊκών κανόνων ανταγωνισμού. Αν κριθεί σκόπιμο να ληφθούν κάποια βήματα και δράσεις, θα γίνει αυτό, ανεξάρτητα από το πότε θα είναι όριμη κατάσταση για μια τέτοια δράση αν παραστεί ανάγκη ανάληψη δράση, αυτή θα αναλυθεί. Αλλά ακόμη δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη. Παίρνουμε στην επόμενη ερώτηση τη κυρία Αντρικιένα με θέμα την προστασία των επενδύσεων στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων Ευρωπαϊκή Ένωση Ρωσία για τη νέα συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. 92 δις ε, των αλλοδαπών ε, παιδίσεων ε, το 2009 ήταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία. Κάτι που την καθιστά το μεγαλύτερο ίσως επενδυτή, αλλοδαπά επενδυτή στη Ρωσία. Σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Είναι πρόθεσή μας να εξασφαλίσουμε ότι οι βασικές αρχές που κατοχυρώνονται στον ενεργειακό χάρτη να αποτελέσουν τμήμα των διαπραγματεύσεών μας με την Ρωσική Ομοσπονδία για τη νέα Συμφωνία Εταιρική Σχέση και Συνεργασία. Οι σχετικέ διατάξει θα πρέπει να, να προβλέπουν προστασία των επενδύσεων στον ενεργειακό κλάδο και ιδιαίτερα έναν ισχυρό μηχανισμό διακαρονισμού των διαφορών. Φυσικά, η νέα αυτή προσέγγιση θα εξαρτηθεί και από τη γενική αξιολόγηση του κατά πόσο ε, ο ενεργειακός χάρτης είναι χρήσιμο πολιτες εργαλείο που θα διέπει τις διεθνεί ενεργειακές σχέσεις. Βασικό του χαρακτηριστικό είναι ότι προβλέπει δεσμευτικούς ε, νομικά κανόνες για την προστασία των επενδύσεων, για την ε, ε, διαμετακόμιση και προβλέπει και κάποιες διατάξεις διακανονισμού των διαφορών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η νέα δέσμευση της Ρωσίας για τη διαδικασία του ενεργειακού χάρτη, όπω φάνηκε στη τελευταία διάσκεψη κορυφής Ευρασίας είναι πολύ σημαντική και η προσέγγιση είναι ανοιχτή και επικοδομητική. Χαιρόμαστε για το ζωηρό ενδιαφέρον της Ρωσίας υπέρ ενός ε, νομικά δεσμευτικού ενεργειακού πλαισίου μετά την πρόσφατη πρόταση για το σχέδιο σύμβασης που θα εξασφαλίσει τη διεθνή ενεργειακή ασφάλεια. Ο εξυγχρονισμός της διαδικασίας του ενεργειακού χάρτη θα είναι το κατάλληλο πλαίσιο για τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις επί της προτάσεως αυτής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Κύριε Αντρικιάννα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Έχω μια συμπληρωματική ερώτηση. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό τον καιρό επεξεργαζόμαστε ε, τη μελλοντική πολιτική επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν μιλούμε για τη Ρωσία, ακούμε συχνά για την επέκταση ρωσικών εταιριών στην ευρωπαϊκή αγορά, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα. Ταυτόχρονα όμως Ευρωπαίοι επενδυτές αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες όταν θέλουν να επενδύσουν στη Ρωσία. Ιδιαίτερα σε κλάδους που θεωρεί στρατηγικούς η Ρωσία, ακριβώς στον ενεργειακό τομέα δηλαδή. Πώς προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει την αρχή της αμοιβαιότητας στις επενδυτικές μας σχέσεις και πώς θα διατηρηθεί αυτό και στη νέα ε, Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης. Ο Επίτροπος. Μάλιστα. Νομίζω την άλλη εβδομάδα θα συναντηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη Ρωσική Κυβέρνηση και θα συζητήσουμε και αυτό το θέμα των επενδύσεων. Εκατέρωθεν έχουμε επιχειρήματα γι' αυτό και η ρωσική πλευρά ε, λέγει ότι ορισμένες από τις δικές της επενδύσεις δεν είναι πάρα πολύ ευπρόσδεκτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί διαρκώς αυτό. Πρέπει να σας πω ότι πέρυσι οι σχέσεις μας γνώρισαν ε, κάποιες δυσκολίες. Τώρα έχουν βελτιωθεί και οι Ρώσοι δείχνουν μεγαλύτερη προθυμία να συζητούν τέτοια θέματα σε βάθος και λεπτομερώς. Ωστόσο, εγώ πιστεύω ότι η εταιρική σχέση και η συνεργασία μας θα βασιστεί στη νέα αυτή συμφωνία και θα πρέπει να έχουμε πολύ ε, μεγάλες ε, ρήτρες προστασίας των επενδύσεων για να αποφύγουμε καταστάσεις ε, τέτοιου τύπου που δεν τηρούν τους κανόνες ε, όλες οι πλευρές. Αυτό είναι μια δυναμική διαδικασία ε, που μας δίνει ελπίδες. Θα υπάρξουν ισχυρές διατάξεις στη νέα συμφωνία γιατί πέρσι υπήρχαν κάποια προβλήματα αλλά τώρα έχει αλλάξει η σχέση μας προς το καλύτερο, θετικότερο. Ερχόμαστε στην επόμενη ερώτηση. η πρόεδρος είναι της κυρίας Γένσεν και αφορά τη στήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Παγκόσμιο Ταμείο για την καταπολέμηση του AIDS, φυματίωση και τη ελονοσίας. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, είναι πολύ εύστοχη η ερώτηση αυτή για ένα θέμα που απασχολεί σοβαρά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς και με μεγάλη ανησυχία και ενδιαφέρον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπέρμαχος ε, του Παγκόσμιου Ταμείου για την καταπολέμηση του AIDS, της κλιματίους και της Ελλονοσία. Ήταν πολύ επιτυχημένη δραστηριότητα αυτού του Ταμείου και στόχος μας είναι να επιλύσουμε τα προβλήματα του Ταμείου το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να συνεχίσουμε να είμαστε οι σημαντικότεροι συνεισφέροντες στο Ταμείο αυτό. Βέβαια, τα προβλήματα που εντοπίσαμε δεν οφείλονται στο ίδιο το Ταμείο, αλλά σε, στον τρόπο που μεμονωμένες χώρες εφαρμόζουν τα προγράμματά του. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις χώρες αυτές ε, για την αποφυγή προβλημάτων κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων. Και μάλιστα ε, το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Παγκόσμιου Ταμείου προέβη σε κάποια έρευνα σε ό,τι αφορά τη χρήση των 4,8 δις ε, δολαρίων σε διάφορες χώρες. Και μάλιστα αυτό γίνεται μετά από καταγγελίες για πιθανές ατασταλίες ή κακοδιαχείριση των κονδυλίων του Ταμείου. Συνεχίζονται και θα ολοκληρωθούν ε, οι έρευνες αυτές. Μάλιστα έχει δημοσιευθεί σχετική έκθεση για το πέρας των ερευνών αυτών στην ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Ταμείου. Οι έρευνες αυτές ήταν ε, διαφανείς και φαίνεται η ε, πολιτική της μηδενικής ανοχής ε, εις βάρος της διαφθοράς εκ μέρους του Ταμείου. Και μάλιστα υπάρχει ένας ε, ανεξάρτητος έλεγχος από το Παγκόσμιο Ταμείο, όπως απαιτείται από τους δημοσιονομικούς κανονισμούς της Ένωσης, για όλους τους οργανισμούς που εποφελούνται από οικονομική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα η έκθεση ελέγχου του 2010 καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το Παγκόσμιο Ταμείο τηρεί και σέβεται τις αρχές του διαχωρισμού των ευθυνών και του ελέγχου διαχείρισης ε, ε, των προγραμμάτων από τις διάφορες χώρες, ώστε οι βασικοί μηχανισμοί και έλεγχοι ισχύουν ώστε τα κονδύλια που λαμβάνουν οι δωρητές ε, να τη χάνουν χρηστής διαχείρισης. Ο ελεκτής βέβαια υπέβαλε πολλές προτάσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης των κονδύλιων, ώστε να απαφευθούν κίνδυνοι κακοδιαχείρισης. Αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξετάζουν ποιες είναι οι δόκιμες τροποποιήσεις προκειμένου να επιταχυθεί η εφαρμογή του προγράμματος του Παγκοσμίου Ταμείου που εγκρίθηκε τον Ιανουάριο και θα γίνει και δεύτερη αποστολή ελέγχου με επισκέψεις σε συγκεκριμένες χώρες για να συνεχιστεί και στην πράξη αυτός ο θεσμικός έλεγχος με επιστολή του Ιανουαρίου του 2011 και μια τηλεδιάσκεψη της Δευτέρας Φεβρουαρίου είχα επαφή με τον εκτελεστικό διευθυντή του Παγκόσμιου Ταμείου, τον κ. Κασέτσκι και του εξέφρασα την επιτακτική ανάγκη περαιτέρω μεταρρυθμίσεων προκειμένου να ενισχυθεί η διαδικασία διαχείρισης του Ταμείου αλλά και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει. Μάλιστα η Γραμματεία του Παγκόσμιου Ταμείου πρότεινε μετά τη τηλεδιάσκεψη την διενέργεια εκτενούς ε, επανεξέταση και να θεωρήσει τον μηχανισμό διαχείρισης. Απαντώντας λοιπόν στην ερώτησή σας κυρία Γένσεν για το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να διακόψει τη χρηματοδότηση στο Παγκόσμιο Ταμείο, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Υπάρχει βέβαια μία αναστολή των πληρωμών, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύω ότι θα πρέπει να τηρήσει τη γενική της δέσμευση προς την υλοποίηση του στόχου του Παγκόσμιου Ταμείου και την ε, ενίσχυση προς τις διάφορες χώρες και τα αισθήματα υγεία τους. Γι' αυτό και προσπαθούμε να θεσπίσουμε συγκεκριμένα κριτήρια που θα πρέπει να εφαρμοστούν πριν προχωρήσουμε σε περαιτέρω συνεισφορές ε, και ξεπάγωμα των ενισχύσεων προς το Παγκόσμιο Ταμείο. Έτσι θα εξασφαλίσουμε και πρόληψη αλλά και σωστή ανείχνευση της απάτης. Κάτι που θα επηρεάσει την ε, δρομολόγηση των προγραμμάτων που ωφελούν τους ασθενείς. Αλλά φυσικά θα πρέπει να ενισχύσουμε τους ελεκτικούς μηχανισμούς και αυτό να γίνει το συντομότερο δυνατό γιατί όσο περνάει ο χρόνος σίγουρα η διακοπή της χρηματοδότησης που ισχύει τώρα δεν είναι η καλύτερη λύση. Χρειαζόμαστε λοιπόν ενισχυμένους ελέγχους σε επίπεδο χώρας ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος κακοδιαχείρισης και να μπορέσουμε να προβούμε στη συνέχιση των πληρωμών. Πάντως, επαναλαμβάνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξακολουθήσει να γίνει σημαντικός δωρητής και ε, συμβάλλον στο Παγκόσμιο Ταμείο, αλλά από τη στιγμή που έχει διαπιστωθεί απάτη θα πρέπει πρώτα να την αντιμετωπίσουμε δεόντως. Πολύ κύριε επίτροπε, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Ε, μόνο τον εισηγητή και ε, δύο θα λάβω, Γένσεν Κάσμαν και μετά ο κύριος Παπα-Νικολάου. Η κυρία Γένσεν, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την ε, υποστήριξή του για το Ταμείο αυτό και επίσης ε, και για το ότι επιθυμεί να παρέμβει σε όλα αυτά τα οποία ε, παρουσιάζουν προβλήματα. Τον ευχαριστώ για το ότι παίρνει σοβαρά το θέμα. Το συγκεκριμένο μου ερώτημα προς τον Επίτροπο είναι το εξής. Τι είδους χρονοδιάγραμμα έχετε κατά νου όσον αφορά το πάγωμα των κονδυλίων του Ταμείου, πόσο γρήγορα μπορεί κανείς ε, να βρει μια λύση. Υπήρξαν συλλήψεις υπόπτων και ε, συνελήφθησαν και οι Εσείς ε, σε πόσο χρονικό διάστημα πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει το θέμα. Ο κύριος Κάσμαν, ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ επίτροπε για την απάντηση συμφωνείτε ότι είναι ζωτική σημασία σε αυτό το Ταμείο Επίτροπε και θα ήταν εγκληματικό να σταματήσει τώρα η χρηματοδότηση γιατί θα τερματιστούν αυτά τα προγράμματα που σώζουν ζωές. Είπατε ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Ταυτόχρονα όμως να ενισχυθεί και η δική μας προσήλωση ε, ότι το Ταμείο αυτό θα βοηθά εκείνους που χρειάζονται περισσότερο ε, τη βοήθειά μας. Ε, για το AIDS, τη και της ελονοσίας και ε, δεν θα πρέπει να πληρώνει αθώοι αυτή τη μάστιγα της διαφθοράς ε, που πλήττονται και απειλούνται από τα τρία αυτά νοσήματα. Ευχαριστώ. κύριος Παπα-Νικολάου παρακαλώ. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την απάντησή σας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση για το Παγκόσμιο Ταμείο σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελαιονοσίας μεταξύ του 2002 και μέχρι το 2010 ε, ε, ε, αφιέρωσε πόρους που ανέρχονται στα 972,5 εκατομμύρια ευρώ που αναλογεί περίπου στο 50% των πόρων του Ταμείου συνολικά. Και ρωτώ, πέραν των όσων μας είπατε για τα προβλήματα που έχετε διαπιστώσει, έχει προβεί η Επιτροπή σε έκθεση αξιολόγησης και σε έρευνα σχετικά με το αν αυτά τα χρήματα πήγαν εξ ολοκλήρου στο στόχο για τον οποίο προορίζονταν. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος, παρακαλώ. Μάλιστα. Δύο είναι τα θέματα εδώ. Αφενός αναγνωρίζω ότι κάνει καταπληκτική δουλειά το Ταμείο ε, και βοηθάει ε, όσους ε, πάσχουν. Δεν χωράει καμιά αμφιβολία. Από την άλλη είναι δημόσιοι πόροι αυτοί και είναι χρήματα των φορολογουμένων. Και έστω και μία περίπτωση διασπάθηση των χρημάτων αυτών μπορεί να καταστρέψει τη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων. Θα πρέπει να βρεθεί λύση το συντομότερο. Μέχρι το καλοκαίρι προτείνω για να επιστρέψουμε σε πληρωμές στο φθινόπωρο. Έχουμε εντοπίσει τους τομείς που χρειάζεται δράση σε επίπεδο κρατών. Γιατί ε, ε το κεντρικό γραφείο έχει ελεγχθεί σωστά. Όταν εμείς θέλουμε τα χρήματα είναι όλα εντάξει, αλλά όταν φτάνουν στους αποδέκτες της χώρες ε, υπάρχει το πρόβλημα. Αν δείτε ποιες χώρες είναι αυτές και τι μέγεθος είχε η χρηματοδότηση, ε, θα ήταν πραγματικά τρομακτικό να μην σταματήσουμε, να μην παγώσουμε πληρωμές. Χρειάζεται άμεση μεταρρυθμίση. Γιατί αν είχαμε ανακαλύψει του χρόνου ατασταλίες, εσείς πρώτοι θα ρωτούσατε, κύριε Επίτροπε, εφού γνωρίζατε την κατάσταση, γιατί δεν αναλάβατε δράση και εγώ θα σας απαντούσα ότι σκέφτομαι μόνο τους ασθενείς και τίποτα άλλο. Όχι, πρέπει να λυθεί το θέμα αυτό. Μέχρι το καλοκαίρι, αν λυθεί στο πρώτο εξάμεινο, δεν νομίζω ε, ότι θα επηρεάσει αυτή η καθυστέρηση ουσιαστικά τη λειτουργία του Ταμείου. Ε, θα έχουμε ενισχύσει όμως την αξιοπιστία του και ε, τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογημένων θα πιάσουν τόπο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Προχωρούμε τώρα στην επόμενη ερώτηση. Ερώτηση προς τον κύριο Ταγιάννη και την έχει υποβάλει ο κύριος Higgins. Θέμα το σήμα CE. So, Commissioner, when you are ready. Κύριε, κυρία Πρόεδρε, ε, αξιότιμε κύριε Higgins, ε, όσον αφορά την σήμανση, αυτό είναι ένα κομμάτι ενός πολύ σημαντικού μηχανισμού για την εύρυθμη λειτουργία της ε, κοινή αγοράς. Η έγκριση του νέου νομοθετικού πλαισίου το 2008 ενισχύει τη διάδοση της σήμανσης ε, με τρεις άξονες. Πρώτον, ε, έλεγχος ε, πιστοποίησης των προϊόντων ΤΣΙΗ. Δεύτερον, έλεγχος των αγορών από πλευράς εθνικών αρχών που οφείλουν να ελέγχουν ε, τη δήλωση ε, συμβατότητας ε, των παραγωγών και των τρίτων κρατών που εισάγουν τα προϊόντα αυτά. Τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να ενισχύσουν τους τελειωνιακούς ελέγχους έτσι ώστε μόνο τα προϊόντα τα οποία σέβονται την νομοθεσία θα πρέπει να κυκλοφορούν. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά εργαλεία για να ελέγξει κανείς στη σήμανση. Τώρα υπάρχει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ενισχύει την αξιοπιστία του σήματος ε, ως εκ τούτου και την ε, καλή φήμη των προϊόντων που παράγονται στην ευρωπαϊκή αγορά και διατίθενται στη διεθνή αγορά. Η ενισχυμένη έλεγχη για τα εισαγόμενα προϊόντα ε, θα οδηγήσουν στο να υπάρχει μικρότερη κατάχρηση του σήματος GS στη διεθνή αγορά. Επειδή λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε σαφές αίτημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιτυχία εφάρμοσε ε, μια, ε, μια εκστρατεία ενημέρωσης ε, σχετικά με το σήμα αυτό εκστρατεία που απευθύνθηκε κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους καταναλωτές. Ο στόχος της εκστρατείας είναι να βοηθηθούν οι ενδιαφερόμενοι κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να κατανοήσουν καλύτερα τη σημασία του σήματος και την λειτουργία του μηχανισμού στον οποίο βασίζεται το σήμα αυτό έτσι ώστε να εφαρμόζονται σωστά οι διατάξεις και να ε, μπορεί κανείς να επερασπιστεί καλύτερα περιπτώσεις παραποίησης προϊόντων ή και επικίνδυνων προϊόντων. Αυτό θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων. Οι συμφωνίες μας με τις τρίτες χώρες συμπεριλαμβανομένων και των χωρών Μερκοσούρου και της Λατινικής Αμερικής κυρίως με την Αργεντινή έχουν ως στόχο να ε, ενισχυθεί περαιτέρω η χρήση του ε, σήματος ΤΣΙΕ. E. Εγώ στις επαφές που θα έχω σκοπεύω να διευκρινίσω τα θέματα αυτά και να προβάλλω τις ε, λύσεις τις οποίες έχουμε καταλήξει. Θα πάω στη Λατινική Αμερική κατά τη διάρκεια της ε, Άνοιξης και το θέμα αυτό λοιπόν θα συμπεριλαμβάνεται στη μερίσια διάταξη των θεμάτων που θα έχω με εκπροσώπους των κρατών που θα επισκεφτώ Βραζιλία, Αργεντινή και Χιλή. Βεβαίως ε, θα ήθελα να επαναλάβω ότι δεσμεύομαι να συνεργαστώ στενά μαζί σας για να υπάρχει σωστή λειτουργία του μηχανισμού που στηρίζει το σήμα GE ε, και επίσης ε, να ληφθούν όλα τα πέντε τα μέτρα για να έχουμε καλύτερη ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας. Προφανώς θα σας κρατώ ενήμερους ε, για τις εξελίξεις και η Επιτροπή μετά από επανέλεγχο της κατάστασης θα παρουσιάσει το 2013 μια νέα εισήγηση της κατάστασης που υπάρχει από το 2008. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Έχω δύο αιτήματα για συμπληρωματική, ο κύριος Χίγγινς πρώτος και μετά η κυρία Τσεκάου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Επίτροπο για την απάντησή του. Είναι πολύ καλή η προσέγγιση με τον καταναλωτή στο κέντρο ε, για προϊόντα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν μπορώ να βρω καμία πληροφορία όμως από πλευρά σας κύριε Επίτροπε, από τη Eurostat ας πούμε, για το τι αξίζει αυτό το σύμβολο για ε, τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και πόσοι οι πολίτες γνωρίζουν τι είναι αυτό το CE. Επίσης θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε περισσότερο. Το 2010, τον Απρίλιο συγκεκριμένα, έγινε μια μεγάλη εκστρατεία ε, σε μια έκθεση στο Ανόβερο ε, για να προβληθεί αυτό το σήμα. Πιάνει τόπο αυτό, τι που έχει κυρία Τσικάου. Ευχαριστώ ε, κύριε πίτροπε. Θα ήθελα ε, να καλωσορίσω τις προσπάθειες που κάνετε για να αναπτυχθεί η βιομηχανική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω σας να ρωτήσω τι ποσοστό των προϊόντων που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέρουν αυτό το σήμα e? και πόσα από τα προϊόντα αυτά παράγονται στην Κίνα και έχουν το σήμα αυτό. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος. Ευχαριστώ πολύ που προβάλλατε ορισμένα προβλήματα που πράγματι βρίσκονται στο κέντρο της προσοχής μας. Γιατί είναι αλήθεια ότι υπάρχει παραποίηση προϊόντων τα οποία εισάγονται νόμιμα ή παράνομα από ε, άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γενικότερα τα κοινωτικά όργανα δεν έχουν τελωνιακούς ε, θεσμούς και δεν έχουν αστυνομικές αρχές ε, που να μας επιτρέπουν να κάνουμε οτιδήποτε άλλο πέρα από το να επαφιόμεθα στις δραστηριότητες των κρατών μελών. Υπάρχουν τα προϊόντα που μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διατίθενται στην αγορά προϊόντα τα οποία πράγματι φέρουν αυτό το εμπορικό σήμα. Εμείς λοιπόν ε, δρομολογήσαμε αυτή την εκστρατεία ενημέρωσης ε, και μετά ε, θα απαντήσω στην άλλη ερώτηση του κυρίου Χίγκινης. Κάναμε λοιπόν αυτή την εκστρατεία όχι μόνο για να χρησιμοποιείται περισσότερο αυτό το εμπορικό σήμα το CE αλλά και για να υπάρχει μια εγγύηση στα προϊόντα και ως εκ τούτου να υπάρχει και μια η χνηλασιμότητα, μια επαλήθευση ε, των παραποιημένων προϊόντων. Στο Ρότερνταμ μπαίνουν πάρα πολλά παιχνίδια. Αυτή είναι μια ιδέα που τη σκέφτομαι ε, και ε, θα πάω και εγώ εκεί προσωπικά στο Ρότερνταμ για να δείξω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για προϊόντα τα οποία εισάγονται από άλλε χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα σε ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια τη Ένωσή μα. Όσον αφορά τώρα τη χρήση του εμπορικού σήματος CE και εγώ νομίζω ότι το σήμα αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται περισσότερο. Ε, βρισκόμαστε στην, σε μια πρώτη φάση και πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, όπως σας είπα, ε, οργανώσαμε αυτή την ενημερωτική εξαρτήση, την οποία συνέβαλε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, θυμάμαι όταν ήμουνα ευρωβουλευτής όλα αυτά που γινόντουσαν τότε που επιμέναμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα σήμα το οποίο θα εγγυάται καταρχήν το σεβασμό των κοινοτικών προδιαγραφών. Γιατί δεν είναι ένα σήμα μόνο ποιότητας ευρωπαϊκής, αλλά είναι και ένα σήμα που ε, εγγυάται ότι έχουν ε, τηρηθεί κάποιες ε, προδιαγραφές, ότι έχουν γίνει σεβαστοί οι κοινοτικοί κανόνες. Γνωρίζω επειδή μου υποβλήθηκε αυτή η ερώτηση και κατά τη διάρκεια της ακρόσης πριν από ένα χρόνο ε, τότε που έθεσα την υποψηφιότητά μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θυμάμαι ότι ορισμένοι βουλευτές είπανε πέρα από το σήμα να περάσουμε και σε ένα... Εγώ προσωπικά δεν είμαι αντίθετο να υπάρχει σήμα, σήμα ευρωπαϊκής ε, ποιότητας. Βεβαίως ε, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να διαδοθεί περισσότερο αυτό το σήμα που υπάρχει, το σήμα και να συνεχίσουμε παράλληλα την ενημερωτική εκστρατεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαφές ότι πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα και μετά σε μια μεταγενέστερη φάση μπορούμε να αρχίσουμε να τα νέες πρωτοβουλίες. Αλλά πριν γίνουν όλα αυτά πιστεύω ότι πρέπει να δουλέψουμε έτσι ώστε το σήμα CE να διαδοθεί περισσότερο σε όλες τις επιχειρήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως στις μικρομεσαίες. Μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες χρειάζονται καλύτερη ενημέρωση. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι εγώ ε, θα συνεχίσω να δουλεύω για να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Higgins ε, που μας προσφέρεται η δυνατότητα μέσα από τη δραστηριότητα των μεμονωμένων ευρωβουλευτών να μιλάμε για τα θέματα αυτά. Μιλάμε και εμείς, οι επίτροποι ε, και ε, τα γραφείο μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με όλα αυτά ενημερώνουμε τα κράτη-μέλη αλλά και τις επιχειρήσεις ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο το είπα και κατά τη διάρκεια της πρώτης μου παρέμβασης, είναι εξίσου σημαντικό να ασκήσουμε πίεση στα κράτη-μέλη για να επαγρυπνούν τόσο στα σύνορα όσο και στο εσωτερικό της αγοράς έτσι ώστε να καταβληθούν προσπάθειες τουλάχιστον να περιοριστεί το φαινόμενο αυτό παραποίησης αυτού του σήματος. Θεωρώ ότι αυτό θα προστατεύσει τα προϊόντα μας αλλά και τους κοινοτικούς κανόνες και όλα αυτά θα είναι τελικά προς του καταναλωτή. Σας ευχαριστώ. Προκειμένου να ικανοποιήσω όλου όσου υπομονετικά περίμεναν στην αίθουσα τη Ολομέλεια, αλλά δεδομένη και τη καθυστέρηση του χρόνου που έχουμε, θα πρότεινα να ομαδοποιήσουμε τις τρεις επόμενε ερωτήσει που είναι αρμοδιότητα του κ. Ταγιάννη και να ακούσουμε τις συμπληρωματικέ ε, από τους τρεις ε, συντάκτες των ερωτήσεων και μετά θα περάσουμε σε ερωτήσεις του κυρίου Σεύκοβιτς. Πρώτη ερώτηση προς τον κύριο Ταγιάννη είναι η ερώτηση Παπα-Νικολάου για το ομοιογενές περιβάλλον ανάπτυξη επιχειρηματικότητα στα κράτη-μέλη. Θα δοθεί απάντηση ταυτόχρονα και στην ερώτηση Κρόλη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην ερώτηση Χάρκιν για την επιχειρηματικότητα στις χώρες που εφαρμόζουν μέτρα λιτότητας. Δεν θέλω να είμαι γενής κυρία Επιτροπέ, αλλά σας θέρμο παρακαλώ να μην ξεπεράσετε, είναι μάλλον να, να τηρήσετε ένα λογικό χρόνο αγόρευσης. θα προσπαθήσω να είμαι σαφής. Θυμάμαι πώς ήταν το πάμε τότε που ήμουν ευρωβουλευτής. Τα θέματα μας είναι πολύ ενδιαφέροντα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πρόθυμη να διατηρήσει το επιχειρηματικό πνεύμα, να βελτιώσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν επιχειρήσεις, κυρίω οι μικρομεσαίες και να τις ενισχύσει έτσι ώστε να έχουν καλύτερη πρόσβαση στις αγορές των τρίτων χωρών. Αυτά τα τρία θέματα είναι προτεραιότητα για, με, για μένα και γι' αυτό το λόγο κατά τις αμέσως επόμενες ημέρες ε, ε, προβλέπω ότι θα γίνει αναθεώρηση του κανονισμού του 2008. Όσον αφορά τις ε, διατάξεις του κανονισμού αυτού, αυτές εντάσσονται στη στρατηγική Ευρώπη του 2020. Όλοι λοιπόν τα κράτη-μέλη θα συμπεριληφθούν σε αυτές τις συζητήσεις και οι επιχειρηματικές οργανώσεις για να ελέγχουμε τα αποτελέσματα. Εμείς σκοπεύουμε να ε, εγγυόμεθα ότι οι αρχές που έχουν ως στόχο να βελτιώσουν την επιχειρηματικότητα ε, θα πρέπει οι αρχές αυτές να εφαρμοστούν τόσο σε κοινωτικό επίπεδο όσο και σε εθνικό. Ήδη έχουμε εισάγει ε, ένα κείμενο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και προσπαθούμε να λάβουμε περισσότερο υπόψη μας τη διαδικασία αξιολόγησης ε, ε, των επιπτώσεων που επηρεάζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στην αναθεώρηση λοιπόν θα υπάρξουν ενέργειες που θα έχουν ως στόχο να βελτιώσουν τις πράξεις μας και να έχουμε καλύτερη αξιολόγηση. Πέρα από αυτό σε όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, εφαρμοστούν οι ίδιες ε, προϋποθέσεις ε, για την εφαρμογή των διατάξεων. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι απαραίτητο να περιοριστεί το διοικητικό άχθος, να υπάρχουν λιγότερες ανομοιογένειες σε εθνικό επίπεδο και ως εκ τούτου θα προτείνουμε συγκεκριμένες δράσεις όπως το One Stop Shop και τις διαδικασίες ε, που ε, υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να έχουμε τις βέλτιστες ε, πρακτικές σε αυτά τα συγκεκριμένα θέματα. Να ενισχύσουμε λοιπόν και το επιχειρηματικό πνεύμα για τους νέους. Πρέπει να βελτιωθούν οι εμπορευματικές κινήσεις και πέρα από τα κοινωτικά σύνορα. Έχουμε το πρόγραμμα Εράσμους για τους νέους επιχειρηματίες και τα αποτελέσματα είναι θετικά. Έχουμε λοιπόν στόχο να εργαστούμε περαιτέρω για να υπάρχει νομοθετική βάση έτσι ώστε αυτό να μετατραπεί σε μόνιμο πιλωτικό πρόγραμμα. Επίση προβλέπουμε παρεμβάσει σε πολύ συγκεκριμένα που αφορούν στις γυναίκε επιχειρηματίε. Έχουμε ένα δίκτυο που σήμερα περιλαμβάνει 250 πρέσβει από 22 χώρες Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω ότι το δίκτυο αυτό μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω. Και τέλο, εργαζόμεθα για να έχουμε προγράμματα προστασία ε, ε, επιχειρηματιών ε, γυναικών σε τουλάχιστον 12 χώρες Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όσον αφορά τη βοήθεια που προσφέρεται μικρομεσαίες επιχειρήσει για τι εξαγωγέ πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις αρχές του περασμένου έτου, ξεκινήσαμε διαβουλεύσει ε, που έχουν ως στόχο το να ενισχυθούν ε, τα μέτρα που υπάρχουν. τα αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων θα μας επιτρέψει να προσαρμόσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές έτσι ώστε να υπάρχουν υπηρεσίες προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και παράλληλα να διασφαλίσουμε τη σωστή χρήση των δημόσιων πόρων. Έχουμε λοιπόν σωρεύσει πολύτιμη εμπειρία ε, όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε προγράμματα ε, που ήταν ε, αποτελεσματικά help desk για την Κίνα, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το κέντρο επιχειρηματικής δραστηριότητας στην στην Ιαπωνία, το Enterprise Europe, ε, το δίκτυο αυτό και πέρα από όλα αυτά ε, με βάση τα αποτελέσματα μιας μελέτης που έχει ανατεθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εκδώσουμε μια ανακοίνωση που θα αφορά στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, στις τρίτες χώρες. Όσον αφορά και κλείνω της αναδυόμενης οικονομίας όπως είναι η Κίνα μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χρησιμοποιήσει τα κονδύλια που έχει εγκρίνει το Κοινοβούλιο έτσι ώστε στην Κίνα και στην Ινδία να υπάρξουν κέντρα παροχής βοήθειας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εγώ προσωπικά ήμουν παρόν τον Νοέμβρη στο Πεκίνο για τα εγγένεια αυτού του κοινοτικού κέντρου ε, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο. Αύριο θα οριστεί ο νέος Mr. Πικ ο Διευθυντής Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ο Γενικός Διευθυντής, ο κύριος Ντανιέλ Καγέχα, ο οποίος θα επιφορτιστεί με το να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς ε, την εφαρμογή των προγραμμάτων και να είναι σημείο αναφορά για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Το έγγραφο που θα εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλούμε όλα τα κρατημέλη να προτείνουν έναν αρμόδιο για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, ο οποίο θα παγρυπνεί για την εφαρμογή της νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να σας πω ότι είχα ήδη θετικές επαφές σε διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, είπα συμπληρωματικέ ερωτήσει από του συντάκτε. Θα ρωτήσω πρωτα πρώτα κύριο Παπα-Νικολάου. Κύριε Επίτροπε, σα ευχαριστώ πολύ για τα όσα είπατε και πράγματι είναι πολύ φιλόδοξα. Ωστόσο, και θα γυρίσω λίγο πίσω το συμβούλιο ανταγωνιστικότητας του δεκεμβρίου του 2008 προσκάλεσε τα κράτη μέλη τότε να μειώσουν το χρόνο εκκίνησης μιας εταιρείας σε τρεις μέρες κατά ανώτατο όριο και η επιτροπή βεβαίως δεσμεύτηκε να παρακολουθήσει αυτή την εξέλιξη τρία χρόνια μετά και μεσούσει τη οικονομική κρίση βλέπουμε στην ελλάδα να χρειάζονται δεκαπέντε μέρε για τη σύσταση μια εταιρεία στην αυστρία έντεκα μέρε στη φιλανδία οκτώ μέρε στο βέλγιο απ' την άλλη μόνο μία μισή μέρα. έχουμε δηλαδή μεγάλε αποκλήσει. και ρωτώ εφόσον η επιχειρηματικότητα συμφωνούμε όλοι ότι είναι προπόθεση για την ανάπτυξη με ποιον τρόπο θα μπορέσει η επιτροπή να περάσει από τι απλέ προτροπέ σε σημαντικέ πιέσει προ κυβερνήσει προκειμένου να μπορέσουμε να εναρμονίσουμε τι διαδικασίε. Ευχαριστώ κύριο Σκρόλη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο και εγώ για την απάντησή του. Τρία σχόλια. Το help desk στην Κίνα. Πολύ ωραία, αλλά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πολύ δύσκολα έχουν πρόσβαση, ιδιαίτερα για τους τομείς που τους ενδιαφέρουν. Φαίνεται ότι βολεύουν περισσότερο τις, μεγάλε τις μεγάλες επιχειρήσεις αυτά τα help desk. Μήπως θα μπορούσαμε καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε στη Βραζιλία, Ινδία, Ρωσία τη συνεργασία και να ενισχύσουμε τις εξαγωγές μας, ενισχύοντας τις επενδύσεις που μπορούν να κάνουν και οι δικές μας επιχειρήσεις. Μέχρι στιγμής το υπόδειγμα ήταν οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιαπωνίας και για το εμπόριο και για τις επενδύσεις και στις δύο πλευρές. αυτό θα πρέπει να είναι το παράδειγμα προς μίμηση και αυτός ο γνώμονας που θα πρέπει να ακολουθήσουμε και για τις σχέσεις με τις άλλες χώρες κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ. Μάλλον θα είναι δύσκολη η ερώτησή μου, γιατί αφορά χώρε που εφαρμόζουν πολύ σοβαρά μέτρα λιτότητα, όπω η πατρίδα μου, η Ιρλανδία. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει χρειάζονται πρόσβαση στην πίστοση, στο δανεισμό. Δυστυχώ δεν τα καταφέρνουν για πολλού και διάφορου λόγου. Γιατί οι τράπεζε θέλουν περισσότερε εγγυήσει από ό,τι μπορούν να παράσχουν οι μικρομεσαίε. Οι μικρομεσαίε δεν θέλουν να αναλάβουν τέτοιο κίνδυνο ε, δανεισμού εκτός από εγγυήσεις των δανείων μπορεί να έχουμε μια πρόταση ίσως για επέκταση του μηχανισμού και του μέσου μικροχρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις μικροπιστώσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που το θέμα των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, για δεύτερη συναπτή ημέρα ε, πυροδοτεί μια κοινοβουλευτική συζήτηση. Εχθές το βράδυ ασχοληθήκαμε με το πώς ε, μπορεί κανείς να διασφαλίσει την πρόσβαση σε κοινοτική χρηματοδότηση ε, τουλάχιστον κατά το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο που θα αφορά στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τι κάναμε και τι κάνουμε για τις επιχειρήσεις αυτές. Όπως σας είπα και κατά διάρκεια της πρώτης μου παρέμβασης και όπως είπα και χτες το βράδυ η βοήθεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για μένα είναι πρώτη προτεραιότητα για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα δεν μπορούμε να μην θεωρούμε αυτό σημαντικό εργαλείο για την έξω από την κρίση. Εργαλείο ενώ τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε την Ευρώπη του 2020 και εκεί βρίσκεται στο επίκεντρό της η πραγματική οικονομία. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, είναι ε, το, η σπονδυλική στήλη, είναι το αίμα αν θέλετε της πραγματική οικονομίας. Και γι' αυτό λοιπόν εγώ πιστεύω και κάτω από το κοινωνικό πρίσμα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να δείξουν καθοριστικό ρόλο γιατί εκείνες θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και αν υπάρξει αναδιάρθρωση ε, των ε, μεγάλων βιομηχανιών. Άρα δηλαδή Πρέπει τις μικρομεσαίες να τις ε, καταστήσουμε ανταγωνιστικές. Ανταγωνιστικότητα σημαίνει καινοτομία και για να είναι κανείς καινοτόμος πρέπει να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στην πίστη. Και αυτό και με τη βοήθεια του Κοινοβουλίου ε, μας οδήγησε στο να έχουμε την απαραίτητη νομοθετική βάση. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό, ε, μια πολύ σημαντική εξέλιξη και ίσως και πριν εκπνεύσει η ε, προθεσμία πλέον ε, θα υπάρχουν διατάξεις που θα ισχύουν για ε, το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 80 περίπου δίσε θα διατεθούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βεβαίως δεν είναι μόνο αυτό. Όπως ανέφερα συντάχθηκε και ένα έγγραφο. Εμείς δώσαμε σάρκα και οστά σε αυτό το έγγραφο για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και στο φόρουμ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ένας νέος ε, θεσμός της Επιτροπής. Εκεί λοιπόν εξετάζονται τα προβλήματα για την πρόσβαση στην πίστη και εκεί εντοπίζονται οι λύσεις για το πρόβλημα αυτό η το χρηματιστήριο του Λονδίνου πίστηκε για πρώτη φορά να συμμετάσχει σε αυτή την πρωτοβουλία και αυτό είναι ένα σημαντικό σημαντικό μήνυμα από τη Μεγάλη Βρετανία είναι ένα μήνυμα υποστήριξης ε, των χρηματοψηφιωτικών κύκλων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βλέπετε λοιπόν ότι και οι κύκλοι αυτοί υποτάσσονται και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην πραγματική οικονομία. Αυτό για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Η δική μου δέσμευση είναι να συνεχίσω να υποστηρίζω την εργασία αυτού του φόρουμ, κυρίως όσον αφορά την πρόσβαση στην δανειοληψία, ε, ε, να υπάρξει κινητικότητα των κεφαλαίων, να μην υπάρχει αυτή η στενοπός ε, που διαφαίνεται αυτή τη στιγμή στο τραπεζικό σύστημα, ε, κυρίως αναφορά τη χρηματοδότηση. Άρα δηλαδή πρέπει να είναι πολύ πιο εύκολη η πρόσβαση στην κοινωτική χρηματοδότηση. Εμείς δουλεύουμε για το επόμενο, το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο, ε, όπως σας είπα λοιπόν και χθε το βράδυ, γιατί δεν ξέρω αν αυτοί που είναι σήμερα εδώ ήταν και χθε παρόντες, όσον αφορά το πρόγραμμα REACH μειώσαμε την φορολογία στο 60% ε, και για τις πολύ μικρές στο 90%. Αυτό λοιπόν τον κανονισμό τον ανέθεσα να ε, μεταφραστεί σε όλες τις κοινωνικές γλώσσες. Αναφέρομαι στην εφαρμογή ε, του προγράμματος REACH. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το ίδιο θα κάνουμε και στον τομέα των κατασκευών. Είχα πολλές συνεδριάσεις για τις μικροπιστώσεις. Πριν από δύο εβδομάδες στις Βρυξέλλες είχαμε μία συνάντηση με τον αρμόδιο της Ιταλικής κυβέρνησης του καινούριου οργανισμού για τις μικροπιστώσεις που νομίζω ότι είναι ένας οργανισμός που λειτουργεί πάρα πολύ καλά και ελπίζω να ενημερωθούμε και για άλλες βέλτιστες πρακτικές από άλλα κρατημέλη έτσι ώστε αυτές να ε, διαδοθούν περαιτέρω όσον αφορά την ανομοιογένεια ε, στους, ε, στις αδειοδοτήσεις αυτό είναι πράγματι ένα πρόβλημα που υπάρχει και γι' αυτό πρέπει να εργαστούμε στα κράτη-μέλη έτσι ώστε να περιοριστεί η γραφειοκρατία Μιλάμε βέβαια για την κοινοτική που έχει τις ευθύνες αλλά υπάρχει και η γραφειοκρατία των ε, κρατών μελών που ανταγωνίζεται αποτελεσματικά αυτή των Βρυξελών. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι όταν λέμε ότι ε, πρέπει να έχουμε κατά νου τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οφείλουμε να μεριμνήσουμε έτσι ώστε και τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν το κείμενο το οποίο έχει αρχίσει να εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επικαιροποιηθεί η νομοθετική βάση και εγώ θα επισκεφθώ τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να δώσω όθηση στα κράτη να ε, χρησιμοποιούν μικρότερα χρονικά διαστήματα, να επιταχύνουν τις ε, διαδικασίες όσον αφορά στι μικρομεσαίε επιχειρήσει, Η Πρόεδρος, ε, συγγνώμη κύριε Επίτροπε, αλλά έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Συγγνώμη και εγώ Πρόεδρε, αλλά το επιχείρημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το όλο θέμα ε, είναι καθοριστική σημασία ε, και γι' αυτό πράγματι μακρηγόρησα περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Σας ζητώ συγγνώμη και από σας προσωπικά και από, τη, από του υπόλοιπου ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ πολύ Επίτροπε. Ερχόμαστε τώρα στι ερωτήσει προ τον Επίτροπο κύριο Σεύκοβιτς. Ελπίζω να έρθει γρήγορα εδώ στο πρώτο έδρανο. Είναι ερώτηση της κυρίας Μπλεκεβιτσούτε με θέμα τη στρατηγική στον τομέα της ισότητας των ευκαιριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Από ό,τι είστε έτοιμος έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που απαντώ τώρα στην ερώτηση αυτή ε, έχω ευχάριστα νέα από την πρώτη πρώτου έχουμε περισσότερες γυναίκες που εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, δεν είναι το τέλος της προσπάθειας. Θα πρέπει να συνεχίσουμε την πολιτική μας να βελτιώσουμε ε, τα στοιχεία γυναικείας παρουσίας ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέσεις διευθυντών και σε θέσεις AD, διοικητικών μη διευθυντών. Στρατηγική 2010-2014 μέχρι την ολοκλήρωση θητείας παρουσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλουμε να έχουμε αποτελέσματα όπου οι γυναίκες θα αντιπροσωπεύουν το 25% της ηγεσίας, 30% στο στα μεσαία στελέχη και 38% των θέσεων AD διοικητικών μη ε, management. Έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των γυναικών το τελευταίο διάστημα. Βεβαίω θέλουμε να συνεχίσουμε τις προσπάθειες αυτές και η μέθοδος που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι ε, αντικατάσταση ε, σε εκείνους που συνταξιοδοτούνται 30% πρόσληψη των ε, ε, γυναικών σε ανώτατες ε, θέσεις και 50% στα μεσαία στελέχη. Δηλαδή οι διευθυντές και οι μάνατζες όταν θα βγαίνουν στη σύνταξη θα αντικαθίσταται από γυναίκες κατά 30% και 50% αντίστοιχα. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχετε καλό μητρό. Τα στοιχεία είναι πολύ εντυπωσιακά. Στο Συμβούλιο δεν ισχύει το ίδιο. Είναι γεγονός ότι κάπως διαφορετικά τα αποτελέσματα αποτελέσματα η καλύτερη μέθοδος είναι για να προχωρήσουμε και να προοδεύσουμε στο μέλλον να συνεχίσουμε την πολιτική μας ανταλλαγής καλών βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουμε τις πολιτικές μας. Ξέρω ότι και οι γενικοί γραμματείς που είναι επικεφαλής των διοικήσεών μας συζητούν αυτό το θέμα σε τακτά χρονικά διαστήματα και αυτή η ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών θα οδηγήσει στα σωστά αποτελέσματα σε όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Μπλίνκεβιτσούτα. Ευχαριστώ. Πολύ καλά νέα και ε, ε, καλωσορίζω και ευχαριστώ για τα όσα μας είπατε για την αύξηση αριθμού γυναικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχω όμως συμπληρωματική ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πόσο καιρό θα χρειαστεί για να ε, μας δηλώσει άλλα ποσοστά, όχι 25% ή 30%, αλλά ακόμα περισσότερα στις ανώτατες διοικητικές θέσεις. Μιλήσατε για το στόχο αυτό και δεν απαντήσατε ακριβώς με μεγάλη σαφήνεια την ερώτησή μου. Ποια είναι η δική σας άποψη, η προσωπική ως επιτρόπου για τη στρατηγική ισότητας ανδρών και γυναικών και οι πιθανότητες που έχουν να καλύπτουν οι γυναίκες ε, υψηλές θέσεις σε όλα τα θεσμικά όργανα και στην ιδιωτική οικονομία. Ε, κυρία Τσεκάου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να διευρύνω κάπως την ερώτηση της προλαλήσης σας και να ρωτήσω τον Επίτροπο αν υπάρχει στρατηγική και για την ισότητα των ευκαιριών των δύο φύλων. Και ενώ εδώ την απασχόληση ε, σε θέσεις ε, διευθυντικές και για επικόους των νέων χωρών μελών. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τις ε, δύο κυρίες για τις συμπληρωματικές ερωτήσεις. Συμφωνώ μαζί σας ότι τα στοιχεία που αναφέρατε μπορεί να, να μην φαίνονται τόσο φιλόδοξα όσο θα προσδοκούσαμε για το μέλλον. Πάντως η αλήθεια είναι ότι όταν ε, ξεκινήσαμε την πολιτική ίσων ευκαιριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1995, έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε έκτοτε την παρουσία των γυναικών στα ανώτατα στελέχη πέντε φορές. Δηλαδή έχουμε πενταπλάσεις ε, θέσεις σε ε, γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις από ό,τι στο παρελθόν. Φυσικά ξεκινήσαμε από πολύ ε, Μέτρια αφετηρία, αλλά θα πρέπει να δούμε και το συνολικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ έρχομαι στη δεύτερη σας ερώτηση. Οι πολιτικές που εφαρμόζουμε για την δημιουργία προϋποθέσεων στις, ε, για την πρόσβαση των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στα κράτη-μέλη, θα πρέπει να βελτιωθούν. Γιατί θα πρέπει να διευκολύνουμε τις γυναίκες ε, με κατάλληλες ε, υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών, με μέρημνας παιδιών, δυνατότητα ελαστικής απασχόλησης, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την ευκολότερη πρόσβαση των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στις χώρες μέλη. Έτσι θα δημιουργήσουμε προδιαγραφέ, ξεκινώντας φυσικά τα θεσμικά όργανα και υπάρχουν πολλά επίπεδα εξασφάλιση τέτοιων ε, θετικών προϋποθέσεων και στα κράτη-μέλη. Με την ε, συνάδελφο Ρέντινγκ προτείνουμε μια στρατηγική για την εξισορρόπηση των φύλων στις ε, ηγετικές διευθυντικές θέσεις επιχειρήσεων και αυτό θα συζητηθεί μέσα σε ένα δίμηνο με επικεφαλής ε, του επιχειρηματικού κόσμου. Δεν ξέρω αν θα επιλέξουμε ένα σύστημα υποχρεωτικών ποσοστώσεων ή θα εφαρμόσουμε το σύστημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή να δημιουργήσουμε πρόσφορες προϋποθέσεις και ενάυσματα στις γενικές διευθύνσεις που πληρούν τους που εκπληρώνουν τους στόχους που έχουμε θέσει για την πρόσβαση των ε, γυναικών. Και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Λυπούμε κύριε Επιτροπή που χρειάστηκε να περιμένετε τόσο πολύ για να απαντήσετε και στο συγγνώμη και από τους διερμηνείς. Οι υπόλοιπε ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν προφορικά θα απαντηθούν γραπτός. Ολοκληρώνεται ο γύρος των ερωτήσεων προς την Επιτροπή και διακόπτεται προσωρινά η σειρά. Ο κύριο Κέλη. Μία παρατήρηση, κυρία Πρόεδρα. Κέλλη, μία παρατήρηση κυρία Πρόεδρε και ξέρω ότι πολλοί συμφωνούν. Δεν έχει καμία σχέση με σας προσωπικά κυρία Πρόεδρε. Είναι θέμα διοργάνωσης των ερωτήσεων. Δεν γνωρίζουμε από την αρχή πόσε ερωτήσει θα απαντηθούν, πόσε συμπληρωματικέ θα υποβληθούν, πόσο θα διαρκέσουν οι απαντήσει και δεν ξέρουμε καν αν ε, θα προλάβει κάποιος επίτροπος απαντήσει στις ερωτήσεις μας. Πραγματικά είμαστε δυσαρεστημένοι. Συνάντησα τη Βαρόνι Λάτφορντ που περίμενε μέχρι τώρα να απαντηθεί η ερώτησή της και άργησε σε ένα δείπνο που ήταν προσκεκλημένη. Εγώ χρειάστηκε να αρνηθώ μια πρόσκληση δείπνου, ελπίζοντα ότι θα απαντηθεί η δική μου ερώτηση. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων πόσε ερωτήσει θα απαντηθούν για να κανονίζουμε και το πρόγραμμά μα. Ξέρω, αλλά αν είναι να λάβουμε γραπτή απάντηση θα μπορούσαμε κάλλιστα από το άνετο σπίτι μας να στέλνουμε ένα mail και να λαμβάνουμε γραπτό στην απάντηση. Δεν έχει καμία σχέση με σας προσωπικά και τον τρόπο διαχείρισης ε, της Προεδρίας, αλλά είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστώ κύριε Κέλλη. Πάντως ως αντιπρόεδρος αρμόδια για την ώρα των ερωτήσεων, με απασχολεί αυτό το θέμα και λυπούμε που ως θεσμικό όργανο δεν καταφέραμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσουμε αυτό που συμφωνήσαμε στη Διοργανική Συμφωνία και να βελτιώσουμε τον τρόπο διεξαγωγής της ώρας των ερωτήσεων. Χαίρομαι που ήρθε ο Επίτροπος Εύτσοβιτς και διαπίστωσε μας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και ελπίζω έτσι ότι θα δημιουργηθεί μια νέα δυναμική και μια νέα όθηση ώστε να υλοποιήσουμε τελικά το στόχο μας ε, όπως ε, συμφωνήθηκε και στη Διοργανική Συμφωνία. ευχαριστώ και πάλι κύριε Κέλλη που θίξατε το ζήτημα. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς και διακόπτουμε τώρα για 7 λεπτά τη σύνοδο μέχρι τις 9 που θα ξαναρχίσουμε.